η διάταξη προχωρούμε στην ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή. Πρώτη ερώτηση κύριου Μπέργκα. Δέκα χρόνια ευρώ. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η εμπειρία που έχουμε από όλο το γενικότερο συντονισμό τα αποτελέσματα θετικά. Όμως θα πρέπει να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. Οι αναλύσεις των πρώτων 10 ετών μας, ε, ε, μας ανεπιβάλλει να συντονίσουμε τις δημοσιονομικές πολιτικές, να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα τα οποία μπορούν να θίξουν τη μακροοικονομική ισορροπία κάποιου κράτους μέλους και την καλή λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία της ε, ΟΝΕ. Αυτός ο καλύτερος συντονισμός θα πρέπει να εξασφαλίσει μια καλύτερη εθνική δημοσιονομική συμπεριφορά και στις καλές στιγμές και στις άσχημες στιγμές. Θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τις, ε, ε, τις εξελίξεις του δημοσίου χρέους και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε εξέλιξη. Ναι, θα πρέπει να έχουμε μια, ένα πιο ενδελεχή μια πιο ενδελεχή δημοσιονομική επίβλεψη, η οποία όμως θα πρέπει να διευρυνθεί για να λάβουμε υπόψη μας και τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ενός κράτους μέλους, παραδείγματος χάρη η, η, η, η αύξηση του, των, των ε, συνεργαματικών ε, αποθεμάτων ε, τάσεις μιας ανισόρροπης εξέλιξης και ανάπτυξης. Η επίβλαψη θα πρέπει βέβαια να στηριχθεί, να στηριχθεί στα ισχύοντα μέτρα και η επίβλεψη και ο συντονισμός προβλέπονται βέβαια στη συνθήκη και στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η πρόσφατη ε, υιοθέτηση του προγράμματος ε, πέρυσι για την οικονομική ανάπτυξη ε, δημιουργεί και μια κάποια επανάσταση αν θέλετε και καινοτομία και εμφανίζει την ρόλο της Κομισιόν αναφορά αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές και την ε, δυνατότητα ε, επιβολής μιας κάποιας σταθερότητας. Η Κομισιόν μπορεί να δώσει μια συγκεκριμένη ε, απάντηση και να δράσει άμεσα σε περίπτωση οικονομικής καθυστέρησης αν θέλετε και στο πρόγραμμα αυτό ανάκαμψης αναφέρονται συγκεκριμένα καθήκοντα. Τα κράτη-μέλη βέβαια είναι υπεύθυνα για τις δημοσιονομικές πολιτικές και η Κομισιόν θέτει έναν γενικό στόχο για περαιτέρω ε, ενθαρρύνσεις, δημοσιονομικές ενθαρρύνσεις έτσι ώστε να ε, δοθεί μια νέα όθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα υπάρχουν νέες προκλήσεις όσον αφορά το συντονισμό και την επίβλεψη της εφαρμογής των νέων ε, μέτρων σε εθνικό επίπεδο. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο Εθνικής Οικονομίας θα ε, παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει το πρόγραμμα ανάκαμψης. Επίσης, ε, η εφαρμογή ε, των ε, μέτρων αυτών που προβλέπονται για την επίβλεψη θα ενδυναμώσει και τις δημοσιονομικές εξελίξεις, θα εφαρμοστούν, θα μπορούν να εφαρμοστούν και καινοτομίε και κάποιες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Βέβαια, δημιουργούνται κάποιες προσδοκίες όσον αφορά την αύξηση του χρέους, αλλά το οποίο θα αντισταθμιστεί από τις ε, περαιτέρω επενδύσεις. Ο κύριος Μπέρκ για μια συγκροματική ερώτηση 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Ε, πραγματικά ευχαριστώ για την απάντηση. Υπάρχει μια κοινή νομισματική πολιτική, αλλά υπό το φως των συνεχιζομένων προβλημάτων θεωρείτε ότι ο ρόλος του Ευρωγκρουπ της Ευρωομάδας θα διευρυνθεί και κυρίως όσον αφορά τις φορολογικές ε, πολιτικές των κρατών μελών και πιστεύετε ότι η υιοθέτηση της συνθήκης της Λισαβόνας θα επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο τις ε, ευρωπαϊκής φορολογίες γιατί το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί πώς μπορούν όλοι αυτοί, αυτά τα νέα μέτρα να ενδυναμώσουν την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη των χωρών της κοινότητας. Κοιτάξτε, ποιος είναι ο ρόλος της, του Eurogroup. Ξέρετε ότι το Eurogroup τώρα και θα συνεχίσει ε, και μετά την υιοθέτηση της συνθήκης της Λισαβόνας μιας μια άτυπη ομάδα. Το, το Eurogroup δεν μπορεί να υιοθετήσει επίσημες αποφάσεις ακόμα και αν αφορά ε, χώρες που ανήκουν στην Ευρωζώνη. Όλες αυτές οι αποφάσεις ε, είναι ευθύνη του Συμβουλίου. Ε, όμως τα τελευταία χρόνια από το καιρό που ανέλαβε την Προεδρία κυρίως ο Ζων Κλοντ Γιούνκερ το 2005 έχει συζητήσει πολλά θέματα και συζητάμε από κοινού με τα μέλη της Eurogroup και με την Κομισιόν και η ACP για την ε, δημοσιονομική επίβλεψη αφενός, αλλά και την ευρύτερη επίβλεψη την οποία ανέφερα. Και στο το Eurogroup συζητάει συχνά και άλλα θέματα τα οποία αφορούν τον εξωτερικό ρόλο του ευρώ και την εξωτερική πτυχή, αν θέλετε, της ε, ε, ζώνης του ευρώ. Οι φορολογίες, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα θέματα και με βάση την τωρινή συμφωνία, αλλά και με βάση την μελλοντική ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Για τις αποφάσεις, ε, για τις φορολογικές, ε, χρειάζεται ομοφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν νομίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα αλλάξει οτιδήποτε σε αυτό το πλαίσιο λήψης αποφάσεων. Έχουμε δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις Επομένως, ο κύριος Λίτφιρτ και μετά ο κύριος Λίνγκριν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψατε μου να σας υποδείξω και να σας τονίσω ότι ε, κάνετε πάρα πολύ τη δουλειά σα, προχωρεί πάρα πολύ καλά η συζήτηση και θα πρέπει να τονίσω στον κύριο Αλμούνια ότι το Eurogroup πάρα πολύ καλά τα πήγε τα τελευταία 10 χρόνια και αυτό το διαπιστώσαμε ω απόδειξη σε αυτή την ε, κρίση. Τόσε χώρε θέλουν να μπουν στο Eurogroup ακριβώ γιατί τι συμφέρει σε αυτέ τι συνθήκε να μπουν σε σχέση με τα σχέδια, εξηγήστε μα, ε, τη Κομισιόν όσον αφορά την μελλοντική σύνδεση του Eurogroup. Δηλαδή τόσε χώρε θέλουν να μπουν μια που έχει αποδείξει το Eurogroup ότι μετράει σαν ε, φορέας. Έχετε το λόγο. Ε, Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Επίτροπο. Μια που ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία του ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια τότε, γιατί η Ιταλία και η Ελλάδα έτσι ενδεικτικά αναφέρω αυτές τις δύο χώρες. Γιατί λέγω αυτές οι δύο χώρες τώρα έχουν χειρότερες επιδόσεις όσον αφορά το δημόσιο χρέος παρότι στο παρελθόν η Σουηδία δε έχει 0,4% χαμηλότερο επιτόκιο από η Γερμανία. Thank you, Madam Μιλάμε για που δεν είναι στο ε, Eurogroup. Ο κ. Σαλμούνια. Όπως ξέρετε πρώτη πρώτου ενό ότο έτου μπήκε η Σλοβαγία στην Ευρωζώνη, οπότε τώρα έχουμε από του 27 16. 16 χώρε οι οποίε τώρα συμμετέχουν. Οπότε όλε αυτέ τι χώρε έχουν το ίδιο νόμισμα και να δούμε τώρα ποιο θα είναι ο επόμενο. Όχι. Δεν απόκειται σε εμά να δώσουμε την απάντηση. Οι υποψήφοι θα ζητήσουν ένταξή τους στην Ευρωζώνη. Βεβαίω. Ε, Πολλέ χώρε θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωζώνη, αλλά δεν πληρώνουν τα κριτήρια τα οποία επιτάσσει η συνθήκη. Οι χώρε τη Βαλτική, η Ουγγαρία και άλλοι. Γνωρίζουμε δε ότι έχουμε δύο κράτη-μέλη την Δανία και τον Ηνωμένο που έχουν αυτοεξαιρεθεί. Οπότε επέλεξαν να μην συμμετάσχουν. Και βέβαια είναι δική τους ε, ευθύνη, δική τους δουλειά το να προετοιμαστούν και κάποια μέρα αν θέλουν να ενταχθούν. Τώρα, ε, ε, Επομένω, μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι μία από αυτέ τι χώρε που έχουν αυτοεξαιρεθεί μπορεί να είναι η πρώτη χώρα που θα μπει στην Ευρωζώνη. σω αυτό γίνεται σε ε, αμέσω στου επόμενου μήνε. σω η Δανία ε, αποφασίσει να μην μετέρχεται αυτή την αυτοεξαίρεση και να ζητήσει να ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Άλλωστε πληρεί όλα τα σχετικά κριτήρια για να μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Όπω ακριβώ τα κριτήρια αυτά τα τάση συνθήκη. Πάση επιπτώσει όμως απόκειται ή στι Δανεικές αρχέ, το Δανέζικο Κοινοβούλιο, ενδεχομένω και στον Δανέζικο λαό τη Δανία, με δημοψήφισμα να αποφασίσουν σχετικώ. Πάντως όπω ξέρετε σήμερα γιορτάσαμε εδώ την δεκάτη επέτειο θέσπιση του ευρώ. Ελπίζουμε ότι κατά την επομένη ετία όλοι, τέλο πάντων σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν ενταχθεί στην Ευρωζώνη, διότι υπό τη σημερινή συγκυρία, υπό αυτού του δύσκολου οικονομικούς καιρού, τα πλέον εκτίματα του να ανήκει κανεί στην Ευρωζώνη είναι ιδιαίτερω υυξημένα για τον παρελθόν. Εκείνοι δε που ακόμη δεν έχουν ενταχθεί, εκείνοι λέγω έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη πιο πολύ το ότι τα πλεονεκτήματα είναι πιο μεγάλα από τις ευθύνες που συνεπάγεται το να ανήκει κανείς στην Ευρωζώνη και τις σχετικές ε, δυσκολίες. Όσον αφορά τώρα τις ε, παρατηρήσεις σας και τις ερωτήσεις σας, εάν ήμουν στη θέση σας, δεν θα έλεγα ότι για το επιτόκια φταίει η Ευρωζώνη. Για ρωτήστε την Δανία. Τι συνέβη με τα επιτόκια. Τι έγινε κατά αυτή την ε, δύσκολη συγκυρία. Μια που η Δανία δεν ανήκει στην Ευρωζώνη. Είδε κεντρική τράπεζα. Ακολούθησε την κεντρική τράπεζα αλλά δεν ε, δεν αντιδρά όσον αφορά αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα υψηλού ρίσκου. Κασάκα. Τώρα όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα και την ε, ευρωπαϊκή αγορά, όσον αφορά την κατάρρευση των τιμών των προϊόντων αυτών. Κύριε Επίτροπε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να εξηγήσω ποια είναι η κατάσταση πριν από μερικά χρόνια. Όλοι θα θυμόσαστε ότι ο λακτοκομικός τομέας ήταν ένας σταθερός τομέας με λίγες διακυμάνσεις στις τιμές. Τα τελευταία χρόνια όμως η κατάσταση άλλαξε άρδινα. Καταρχάς το 2007, από ό,τι θυμάμαι, θυμάμαι και πάρα πολύ ε, καλά, το Σεπτέμβριο του 2007 είχαμε σημαντικές αυξήσεις στην τιμή των γαλακτοκομικών προϊόντων και μετά πέρσι είχαμε μείωση σημαντικότητα στις τιμές. Επομένως η κατάσταση είναι ότι οι τιμές προσεγγίζουν τις τιμές παρέμβασης και σε ορισμένες χώρες έχουν κατέβει κάτω και από το κατόφλι αυτό των τιμών παρέμβασης. Ξέρω ότι θα πρέπει να, να, να σας πω ότι με ανησυχεί ιδιαίτερα η επιδείνωση του γαλακτοκομικού τομέα και της αγοράς των γαλακτοκομικών προϊόντων. Έχουμε μέτρα υποστήριξης, τα οποία εφαρμόζουμε, που ήδη έχουν ξεκινήσει να υποστηρίζουν το γαλακτοκομικό τομέα και έχουμε αναλάβει δράση ήδη. Αντίθετα από την κανονική ε, κατάσταση όπου τα συστήματα για την αποθεματοποίηση του βουτύρου ξεκινάνε από την 1η Μαρτίου. Εμείς προτείνουμε από την 1η Ιανουαρίου να ξεκινήσει ε, το μέτρο αυτό, έτσι ώστε η παραγωγή του Δεκεμβρίου να είναι επιλέξιμη για το μέτρο αυτό οι αγορές στην παρέμβαση ή η χορήγηση εξαγωγικών επιστροφών είναι άλλα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τον γαλακτοκομικό τομέα αποτελεσματικά. Όσον αφορά τώρα το σύστημα παρέμβασης που ξεκινάει τον Μάρτιο και που καλύπτει και την παραγωγή η οποία θα λάβει χώρο τον Φεβρουάριο για το βούτυρο και για το αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη μπορούν να αγοραστούν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Και για τις σταθερές ποσότητες που θα είναι σε σταθερές τιμές και μετά θα υπάρχει η, η διακύμανση που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και ποια είναι η κατάσταση που επικρατούσε το 2007. Θα θυμόσαστε όλοι την άμεση ε, απάντηση που εδόθη από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από το Συμβούλιο, από τα κράτη-μέλη με πιέσατε ιδιαίτερα να αυξήσω άμεσα, ή από χτες ας πούμε και όχι σήμερα ή αύριο, να αυξήσω τις ποσοστώσεις, να χαλαρώσουμε λίγο την κατάσταση όσον αφορά τις τιμές του καταναλωτή. Και θα ήθελα επίσης να μιλήσω ξεκάθαρα σήμερα για να ε, μην υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας ότι η αύξηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων ε, θα πρέπει να θεωρηθούν οι υπεύθυνε για την ε, επιδείνωση της αγοράς. Η πραγματικότητα είναι ότι παρά την αύξηση κατά 2% των ποσοστώσεων που έλαβε χώρα τον Απρίλιο πέρυσι, η μείωση υπήρξε μείωση της παραγωγής, διότι η παραγωγή, η αύξηση των ποσοστώσεων παρουσιάζει μια δυνατότητα για τα κράτη-μέλη και για τους αγρότες να, να παράγουν περισσότερο, αλλά δεν είναι υποχρέωση. Επομένως βλέπουμε ότι η παραγωγή ε, και οι καταναλωτές ε, απαντούν στα, στις ενδείξεις της αγοράς οι αλλαγές, οι μικρές αυτές αλλαγές που είδαμε στο σύστημα των ποσοστώσεων δεν εξηγούν κατά έναν τρόπο την ε, διακύμαση στην αγορά και την αστάθεια της αγοράς. Η μη χαμηλή ε, ζήτηση από πλευρά των καταναλωτών είναι ίσως ένα αποτέλεσμα της, ε, των υψηλών τιμών που είχαμε πέρυσι, διότι οι καταναλωτές δεν αγόρασαν τα πολύ ακριβά γαλακτοκομικά προϊόντα και ίσως αυτή να είναι, αυτός είναι ο λόγος για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Επομένως, ε, δεν θα πρέπει όμως να ε, βαφκαλιζόμαστε ότι κάνοντας μικροαλλαγές στον γαλακτοκομικό τομέα ε, μπορούμε να επηρεάσουμε το, στο σύνολο του τομέα. Άρα το ποσοστό ε, ε, συγγνώμη, το, η αλλαγή στο σύστημα των ποσοστώσεων δεν άλλαξε και δεν σταθεροποίησε την ε, αγορά. Τώρα, οι πορτογαλικές αρχές χρησιμοποίησαν κάθε δυνατότητα για την αύξηση, για να ζητήσουν την αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής γάλακτος για τα νησιά. Και οι Αζόρες, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ε, εποφελούνται από την αύξηση της παραγωγής, από τη δυνατότητα αύξηση της παραγωγής. Είναι σε προνομιακή θέση. Και είμαι σίγουρη ότι οι μεγαλύτερες ποσοστώσεις θα είναι προς όφελος της γαλακτοκομικής παραγωγής της Αζόρες. Και τα νησιά αυτά είναι αρκετά απομακρυσμένα και θα πρέπει ανάμεσα στα νησιά αυτά να γίνεται και η μεταφορά του γάλακτος. Για να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, να διαβεβαιώσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θα διαχειριστώ την, τα εργαλεία που μας παρουσιάζει, που μας διαθέτει η πολιτική μας στο γαλακτοκομικό τομέα, έτσι ώστε να δημιουργήσω ένα δίκτυο ασφάλειας για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ο κύριος Καζάκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο. Επίτροπε. Αλλά κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ με την αισιοδοξία σας για τον τρόπο ε, η αύξηση, οι αυξήσεις των ποσοστώσεων θα είναι προς όφελος των αζωρών να σας πω κυρία Επίτροπε ότι έχουν γίνει κάποιες αξιολογήσεις και, κάποιες, και έχουμε κάτα, και κάποια στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευθεί και μιλούν για μείωση των τιμών σε γάλα σε σκόνη που θα θίξουν ε, τις, ε, τα εισοδήματα των αγροτών όχι μόνο στις Αζόρες αλλά και αλλού. Και αυτές οι διατάξεις, αυτά τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν δεν είχαν καμία συνέπεια και κανένα αντίκτυπο στην ε, περιοχή μου. Η κυρία Επίτροπος θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Thank you. Ε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ξέρετε ότι πάντοτε με χαρά συμμετέχω σε διάλογο και συζητήσεις μαζί σας για τη σημασία του τομέα της γεωργίας και ιδιαίτερα για τις αζόρες. Βρισκόμαστε πιστεύω σε μια ιδιαίτερη κατάσταση σήμερα. Η αγορά δηλαδή αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες. Είναι πολύ δύσκολη και αυτό ισχύει όχι μόνο για τις Αζόρες αλλά γενικότερα για την Ευρώπη ολόκληρη. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι τιμές έχουν πέσει σε επίπεδο αδιανόητο μέχρι πριν από, τρεις, από έξι μήνες. και σας διαβεβαιώ, φαντάζομαι ότι θα γνωρίζετε, θα πιστεύετε κι εσείς ως συνήθως, πως θα μπορέσω να βρω τις κατάλληλες λύσεις. Αυτή είναι η προσπάθειά μου και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπό τις συγκεκριμένε συνθήκες. Κυρία Μαγκίνες, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλή χρονιά, Επιτροπή. Και ας μην είναι καλά τα νέα για τα γαλακτοκομικά μας. Είπατε, αναφερθήκατε σε κάποιους από τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά, αλλά μια και κάποια θέματα δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρα ως προς την ε, πτώση αυτή τη δραστική των τιμών. Έχετε βεβαιότητα, όταν τα πάντα και οι πάντε είναι αβέβαιοι για την κατάσταση. Έχετε βεβαιότητα ότι τα μέτρα αυτά θα μπορέσουν να βοηθήσουν και ότι θα αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη αυτή που θα βοηθούσε στο να αντιμετωπιστεί αυτή η πτώση στην παραγωγή, ακόμη και στην παραγωγή, η μείωση τη παραγωγή. υπάρχουν διάφοροι λόγοι που εμφανίζεται αυτή η κακή παραγωγή γάλακτος. Κύριος λόγος είναι η τεράστια σημασία της ρωσικής αγοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία τώρα στην οικονομία της, όπως βλέπουμε πρόσφατα, αντιμετωπίζει μια τεράστια υποτίμηση Επομένως ε, υποβαθμίζεται σημαντικά η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Έχουμε, δεν έχω ακριβή στοιχεία, αλλά έχουμε τουλάχιστον 15% ε, υποτίμηση, άρα μειώνεται σημαντικά η δυνατότητά μας να πωλήσουμε προϊόντα στη Ρωσία. Συνέπεια των υψηλών τιμών που είδαμε το 2007, εξάλλου, είναι να αποφεύγει ο κόσμος τα πιο ακριβά γαλακτοκομικά από τότε μέχρι τώρα, ακόμα δεν έχει αναστραφεί αυτή η τάση και βέβαια και η αβεβαιότητα εντωμεταξύ λόγω της γενικότερη οικονομικής κατάστασης. Επίσης η κύριε Μακίνες ρωτάει εάν θεωρεί ότι το check-up για τη γεωργία αρκεί μετά όσα κάναμε εκεί. Κοιτάξτε, το check-up δεν ξεκινάει πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2010 και όλα τα μέσα που έχουμε στη θέσή μα για του διαφορου τομεί ξεχωριστά θα αρχίσουν να λειτουργούν από τότε. Βλέπουμε λοιπόν και το βλέπουμε από τι συζητήσει ότι έχουμε μπροστά μα και νέε προκλήσει. και μπορούμε να διαθέσουμε διαβαθμισμένα τα χρήματα για τι νέε αυτέ προκλήσεις αλλά όχι για το 2009, δεν είναι διαθέσιμα αυτά ποσά. Και γι' αυτό προτείνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βέβαια, στο ΕΚΟΦΗΝ, κάποια από τα μη απορροφηθέντα κονδύλια, 5 δίσεν από την ε, γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου, 1,5 δις συγκεκριμένα από την ανάπτυξη της υπαίθρου, να δαπανηθούν τώρα, το 2009. Το Κοινοβούλιο από εκεί και πέρα και το Συμβούλιο έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την απόφαση εάν είναι δυνατόν να δαπανηθούν κάποια από τα χρήματα αυτά. Αν θυμάστε το κατάλογο των νέων προκλήσεων, συμπεριλαμβάνε και τον τομέα των γαλακτοκομικών. Και ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια κατανόηση και από πλευρά του Κοινοβουλίου, έτσι τα χρήματα αυτά να δαπανηθούν και, όχι αποκλειστικά, και για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίσουν το πνεύμα των γαλακτοκομικών. Μικροπιστώσει. Βαν Χέκε, έχει υποβάλει την ερώτηση. Ε, είναι μια ερώτηση που απευθύνεται προ τον Επίτροπο, τον κύριο Μισελ. Κύριε Άλιστερ, έχετε το λόγο. μετά από μία ερώτηση. Δεν δέχεστε δύο συμπληρωματικέ, δεν ρώτησα εγώ το λόγο και δεν είπα προ την Επίτροπο ε, ότι έχω μία συμπληρωματική, γιατί δεν μου δώσε το λόγο για την συμπληρωματική, Πρόεδρο. Δεν το κατάλαβα ότι το ζητήσατε αυτό, κύριε Αλιστερ. Αν το καταλάβαινα, φυσικά και θα σα έδινα το λόγο. Άλιστερ. Μα οι καθήμενοι δίπλα σα το, το προσωπικό κοινοβουλίο, είπαν ότι ελήφθη υπόψη το ότι ζήτησα το λόγο. Άρα, γιατί δεν σα το είπαν. Γιατί δεν το ξέρατε. Όχι, όχι, όχι. Από ό,τι μου λένε και μου επιβεβαιώνουν, δεν σα είδαν. Κύριε Μισελ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι οι επαφές Συμβουλίου και Επιτροπής αποσκοπούσαν στο να έχουμε κάποιον κανονισμό και είπαμε να μην χρησιμοποιήσουμε αυτό το οποίο επιτρέπει το κεφάλαιο 2 του προπολογισμού. Αντίθετα με τις προτάσεις της Επιτροπής. Οπότε ο κανονισμός της 16ης Δεκεμβρίου του 2008 προβλέπει ένα δις από το τέταρτο κεφάλαιο. Αυτό θα χρηματοδοτήσει την περίοδο από το 2008 έως το 2010 θα χρηματοδοτήσει κάποια μέτρα στήριξης της γεωργίας και της ε, διατροφικής ασφάλειας όσον αφορά την κάλυψη της ε, διατροφικής κρίσης. Οι δε μικροαπιστέσεις ε, εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτά τα μέτρα. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε την αύξηση της παραγωγής. Έχουμε κάποιες τέτοιες δράσεις χρηματοπιστωτικές για τέτοιες διευκολύνσεις, κάτι το οποίο γίνεται πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, γίνεται με την διαδικασία της Επιτροπολογίας όσο προβλέπετε και έχουμε ένα πρώτο πακέτο 300 εκατομμύριων ευρώ και αφορά 25 χώρες. Ε, θα παρουσιαστεί αυτό μας το πρόγραμμα τον ε, Φεβρουάριο. Ε, επίσης θα προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί το σύνολο αυτής της διευκόλυνσης, κάτι το οποίο θέλουμε να ψηφιστεί πριν την 1η Μαΐου 2009. Εμείς είμαστε υπέρ του να αναπτυχθεί αυτό το μέσο των μικροπιστώσεων ε, και γενικά της μικροχρηματοδότησης. Οπότε έτσι έχουμε ε, όλη αυτή τη βεντάλια μέτρων με μεταφορά πόρων και συστήματα ε, πληρωμών. Εμείς έχουμε δεσμευθεί τους ε, λιγότερο προνομίχους να τους βοηθήσουμε ούτως ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες ε, υπηρεσίες χρηματοδότησης γιατί υπάρχουν προβλήματα, προβλήματα όσον αφορά τις, τεχνικές. Τα χρήματα όμως υπάρχουν, άρα θα πρέπει να αρθούν αυτοί οι φραγμοί και να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και κυρίως δηλαδή να χρησιμοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες αυτοί που τις έχουν ανάγκη. Γι' αυτό και εμείς επικεντρώνουμε προσπαθειές μας όσον αφορά την ενίσχυση των θεσμικών δυνατοτήτων που αφορούν τις μικροπιστώσεις και όσον αφορά την πρόσβαση στο κεφάλαιο είναι τόσο σημαντική για τις μικροπιστώσεις ας πούμε εκεί όπου έχουμε μικροχρηματοδότηση σε κάποια ζώνη της υπαίθρου εμείς πρόκειται να καλύψουμε τις χρηματοπιστωτικές ανάγκες μέσω Κάποιε τράπεζες εξειδικευμένε όπω η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρησιμοποιώντα τι πιστώσει, τους ώστε να μπορεί κανεί να πάρει κάποιο δάνειο, να έχει και κάλυψη ε, ακόμα και αν χρειαστεί να έχουμε ε, startup, κάποιο καινούριο ε, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Θα βοηθήσουν και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, θα έχουμε έτσι συγκριτικό πλεονέκτημα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαχειρίζεται αυτέ τι ε, τις, τις, τις δράσεις μικροχρηματοδότησης. Για δε την ε, ε, Μεσόγειο έχουμε το FMP και έτσι ε, μπορούμε να καλύψουμε ότι ακόμα και χώρες της ΑΚΕ. Ο κ. Βαν χέκια τώρα έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου. Μικρό. Νάψε το μικρόφωνο σας λέει ο Πρόεδρος. Η απόφαση να αποδεσμευθούν τα ποσά, τα ποσά αυτά για τις, ε, προς των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση είναι ένα μέτρο το οποίο υποστηρίξαμε όλοι μας. Η Κομισιόν όμως πρότεινε υπό την πίεση κάποιων κρατών, κρατών και από ένα μέρος του Κοινοβουλίου να χρησιμοποιήσει τους πόρους που δεν χρησιμοποιήθηκαν γιατί είναι γεωργία. Πιστεύετε ότι η χρήση αυτών των πόρων ε, θα είναι χρήσιμη για την καταπολέμηση της φτώχειας. Μιλήσαμε για την προσβασιμότητα. Είπαμε ότι είναι ένα μέτρο για τις πόλεις, όχι για την Ήπεθρο. Και η ερώτηση προς την Κομισιόν έγινε μια γενική αξιολόγηση του εργαλείου αυτού. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, προετοιμάζουμε τον μηχανισμό ο οποίος θα επιτρέψει να εφαρμόσουμε άμεσα και να χορηγήσουμε τα δημοσιονομικά, τα οικονομικά ποσά, τα οποία, τα ποσά μάλλον, τα οποία ε, έχουμε αποφασίσει, όμως η φύση ή η προέλευση των πόρων μα δεν μας δημιουργεί πρόβλημα. Ακόμα και στην περίπτωση ε, project που αφορούν την Ήπεθρο, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση, δεν έχουμε καμία δυσκολία. Σας καθησυχάζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και ούτως ή άλλως θα, λάβουμε υπόψη μας την ανησυχία που εκφράσατε, θα το δείτε στο πρώτο πακέτο το οποίο θα υποβληθεί τέλος Φεβρουαρίου ή και στο γενικότερο πλαίσιο το οποίο θα ε, είναι έτοιμο έτοιμο για την 1η Μαΐου. Κύριος Λίμπφιλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Μια σύντομη ερώτηση. Υπάρχει πρόθεση, έχει κανείς αναλογιστεί τη δυνατότητα να προβλεφθούν συγκεκριμένοι στόχοι και να οριστούν ανώτατα επίπεδα συγκεντρώσεων ως προς τα τρόφιμα κτλ. Υπάρχει κάτι εδώ. Κύριε Πίτροπε. Φυσικά, η απάντηση. Δεν μπορώ να περάσω στην διαχείριση των αναπτυσσόμενων κρατών και να την σχολιάσω εγώ. Είναι γενικά πολύ ευάλωτες δομές. Αυτό που προτείνετε εσείς ως ερώτηση υποθέτω ότι υπονοεί κάποια συγκεκριμένη κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμό. Βλέπω ότι εννοείται και μου φαίνεται αρκετά κατανοητό και θετικό εκ πρώτης όψεως. Πρόκειται για μια ερώτηση θα μπορούσα να ενσωματώσω στις συζητήσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή και να επανέλθω για να δούμε πώς μπορούμε να οργανωθούμε. Φαντάζομαι ότι εννοείται κίνητρα τα οποία θα μπορούσαν να ε, δώσουν να καθοδηγήσουν περισσότερο προς την οικογενειακή βιοτεχνική γεωργία, τη λεγόμενη και βιολογική αν θέλετε, που θα μπορούσαμε βεβαίω ναι, να αναζητήσουμε ε, εφόσον βέβαια υπάρχει και δυνατότητα να έχουμε και τη σχετική διάθεση στον ευρύτερο χώρο. Γιατί έχουμε μια χώρα με μεγαλύτερη παραγωγή από ό,τι χρειάζεται, χρειάζεται βέβαια η διαφοροποίηση. Πολύ ευχαρίστω ε, να το διερευνήσουν. Χρήσιμη η υπόδειξή σας και θα την ε, μεταφέρω στις υπηρεσίες μου, να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το ενσωματώσουμε στα σχέδιά μας. Mm. Κυρία Μαγκίνες και παρακαλώ να είναι σύντομη διότι έχουμε καθυστερήσει. Ναι, όντως ήθελα να ρωτήσω για τα... Για... Ήθελα να ξέρω μήπως λόγω της οικονομικής κρίσης η Κομισιό έχει υποβαθμίσει λίγο στην ημερήσια διάταξή της τα θέματα της παγκόσμιας ε, ε, επιστηστικής ασφάλειας διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, τα παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από την πείνα. Κοιτάξτε, αυτό δεν, είναι, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν συζητάμε κάθε μέρα ε, κάποια θέματα δεν μας απασχολούν και δεν ε, ασχολούμεθα μαζί τους. Η Κομισιόν συνεχίζει τις εργασίες που έχει ξεκινήσει ήδη με την βοήθεια του Κοινοβουλίου. Σας θα ήθελα να σας καθησυχάσω. Ε, και να σας πω επίσης ότι το θέμα είναι ενδιαφέρον, η ερώτησή σας ήταν ενδιαφέρουσα, διότι το γεγονός ότι μείωσ... μειώθηκαν οι τιμές ε, λόγω της ε, ε, κρίσης θα, μπορούσαν, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι λύθη έχει επιληθεί και το πρόβλημα. Όχι, μπορεί να μειώθηκαν οι τιμές αλλά δεν έχουμε φτάσει στο χαμηλό επίπεδο το οποίο ισχύει στο παρελθόν και η, η διατροφική αν θέλετε κρίση θα συνεχίσει να είναι πρόβλημα και τα επόμενα χρόνια. Επομένως θα επαγρυπνούμε, μην ανησυχείτε, δεν ξεχνάμε το θέμα αυτό διατροφικής ασφάλειας. Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο τμήμα. Καταρχάς, ερώτηση της κυρίας Άρκιν για την ε, μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού. Κυρία Γκριμπαουσκάιτε, έχει το λόγο. Δύο ερωτήσεις έχουμε για την ομόρφωση του προπολογισμού. Η μία αφορά ειδικότερα τα θέματα ε, τα γεωργικά. Ζήτεται να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτά τα θέματα. Η πρώτη ερώτηση, όπως είπα, είναι γενικότερη υφής, ε, αφορά την αποτελεσματικότητα του προϋπολογισμού. Έχουμε δημόσιες ε, διαβουλεύσεις, επικεντρώθηκαν στο πώς ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα είναι πιο αποτελεσματικός, πιο απλός, με περισσότερη διαφάνεια. Αυτό πρόκειψε από την διαβούλευση που έγινε. Ζητείτε απλούστευση και αναλογικότης όσον αφορά τα διοικητικά αλλά και τον έλεγχο. Επισημάθηκαν κάποια δυνατά σημεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έλαβε υπόψη πολλά από αυτά τα σχόλια και ήδη έχουμε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια και έτσι αντιδράσαμε για να έχουμε περισσότερη προσβασιμότητα και πιο ανοιχτό πνεύμα στον αφορά τον προπολογισμό. Επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρότητα με κάποια σημεία τα οποία ανέγυψαν από την δημοσία διαβούλευση πρώτα-πρώτα όσον αφορά την εσωτερήκευση κάποιων δαπανών. Δηλαδή το, αυτό που ονομάζεται ε, ένταξη στον προϋπολογισμό, ε, νομιμοποίηση αυτών των δαπανών ούτως υπήν μέσω της ένταξης στον προϋπολογισμό. Ο, βέβαια ακόμα δεν ολοκληρώθηκε το έργο μας ε, σε αυτό το σημείο. Επίσης και το έργο των κρατών μελών είναι κρίσιμο. Και έτσι θα πρέπει να λάβετε υπόψη το ότι σε πάρα πολλούς τομείς διαχειρίζονται κράτη-μέλη 80%. Θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ αυστηρή οριοθέτηση των αρμοδίτων κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι το οποίο θα επιτευχθεί όταν ισχύσει η συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Τώρα, όσον αφορά την έλλειψη ευελιξίας εκ του προπολογισμού ε, πρόσφατα, όσον αφορά τις διευκολύνσεις για την διατροφή, ε, όσον αφορά την κρίση με το φυσικό αέριο όσον αφορά την ε, ανασυγκρότηση τη της ευρωπαϊκής οικονομίας φάνηκε το ότι ο προπολογισμό δεν έχει την αναγκαία ευελιξία. Οπότε φάνηκε ότι θα πρέπει εκεί να επενδύσουμε στις λειτουργικές δυνατότητες αντίδρασης του προπολογισμού. Άλλα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν κατά την διαβούλευση αφορούν την ελαχιστοποίηση των διοικητικών δαπανών. Ήδη έχουμε δεσμευθεί σχετικώς, έχουμε αναλάβει και κάποιο πρόγραμμα δράσης που περιλαμβάνει και εσωτερικούς ελέγχους. Απλούστευση επίσης των διατάξεων όσον αφορά διάφορες διατάξεις. Όσον αφορά κάποια εφάπαξ ποσά, ε, κάποιες πληρωμές που προβλέπονται. Οπότε θα πρέπει τώρα να επανακαθορίσουμε το σύστημα ελέγχου όσον αφορά τα επίπεδα αποδεκτού λάθους και, τους, και την ισορροπία κόστους κινδύνου. Συμφωνούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την, τον εξορθολογισμό και απλούστευση του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ για την ερώτηση που υποβάλλατε. Ξέρω ότι δεν είναι τόσο συναρπαστικό το θέμα, θεωρείται υπερβαλλόντος τεχνικό, αλλά ό,τι πολιτικές αποφάσεις και εάν δεν έχουμε αποτελεσματικό προπολογισμό, μια σωστή πολιτική δεν θα πιάσει τόπο. Η Πρόεδρος. Ήδη έχουμε καθυστερήσει σημαντικά. Άρα θα πρέπει τις συλλογικές οτήσεις να τις ομαδοποιήσουμε. Κυρία Χάρκιν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που απαντήσατε σε όλα μαζί είπατε για ευθύνες των κρατών μελών. Μπορείτε να μας συγκεκριμενοποιήσετε τι γίνεται όσον αφορά το κόστος της επιλεξιμότητας, τι γίνεται με αυτές τις εφάπαξ πληρωμές, τι γίνεται με τα διευθυντικά ταμεία, τι γίνεται με αυτό το έγγραφο της διαβούλευσης, τι γίνεται με τη Γεωργία. Αν ρίξει μια ματιά κανείς το τι προέκυψε, λέει για ποικιλία, ε, γνώση, ε, αλλαγή κλίματος, ενέργεια. Δεν λέτε πουθενά στην, ε, στο έγγραφο αυτό της διαβούλευσης για διατροφική ασφάλεια. Πόσο έχετε επηρεαστεί από αυτό το έγγραφο. Κυρία Πίτρο, μισό λεπτό να υποβάλουμε τις ερωτήσεις όλες μαζί. Η κυρία Τικά, όχι το λόγο παρακαλώ, σεβαστείτε το χρονικό όριο γιατί έχουμε καθυστερήσει πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, στα ρουμανικά. Θα ήθελα να σας πω ότι η χρήση 2009 είναι η χρονιά της καινοτομία και της δημιουργικότητας, οπότε έχουμε όμως και μια άλλη προτεραιότητα, την αλλαγή του κλίματος. Να μην ξεχνούμε δε ότι όσον αφορά το πρόγραμμα της ανασυγκρότησης της, ε, και αναθέρμανσης οικονομίας, θα πρέπει να δοθεί στα έργα υποδομής προτεραιότητα για μεταφορά και ενέργεια. Αυτές είναι προτεραιότητες. Πώς αυτά θα τα εντάξετε στη μεταρρύθμιση του προπολογισμού. Η Επίτροπος έχει το λόγο. Mm. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τρεις συμπληρωματικές ερωτήσεις για τα τα ταμεία, η πρώτη και το τι έχουμε κάνει. Εμείς ε, διαπραγματευόμαστε ε, με το Κοινοβούλιο για, τις, ε, για το δημοσιονομικό, δημοσιονομικές προοπτικές τέλος πάντων και για τον προπολογισμό και θέλουμε να είναι πιο ευέλικτο το σύστημα που, ε, που θα εφαρμόζεται για τα κράτη-μέλη κυρίως όσον αφορά την, ε, και τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και το πρόγραμμα, ε, το σχέδιο ανάκαμψης. 6 δισεκατομμύρια έχουμε αναλάβει υποχρέωση απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα διαρθρωτικά ταμεία και τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο υποστήριξαν την πρόταση αυτή. Ε, ήδη έχουν γίνει κάποιες προτάσεις για την αλλαγή των κανονισμών και νομίζω ότι ε, και για την ε, περιφερειακή πολιτική και θα περάσουν και από το Κοινοβούλιο. Τώρα, όσον αφορά την διατροφική ασφάλεια, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα γενικώ για την κοινή γεωργική πολιτική εν γέννη. Και το πρόβλημα είναι η ποιότητα της κοινής γεωργικής πολιτικής, η δυνατότητα να αντιδράσει και να βοηθήσει. Οι πολιτικές είναι αρκετά δαπανηρές και το συνειδητοποιούν αυτό οι συμμετέχοντες στην πολιτική αυτή. Όντως η πολιτική αυτή στο άμεσο μέλλον και με, μέσω πρόθεσμα ε, δεν θα, μάλλον θα ε, επενδύει περισσότερο σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας της υγείας. Ε, έτσι βλέπουμε εμείς το πρόθεσμο μέλλον. Δεν μπορούν όμως όλοι να το δούνε αυτό. Προσπαθούμε να είμαστε αντικειμενικοί ε, δημοσιεύουμε όλο το υλικό μας και όλες τις πληροφορίες που έχουμε. Όλα δημοσιεύονται. και τη σύνοψη και τις διαπραγματεύσεις μας. Επομένως, Προσπαθούμε, προσπαθούμε να είμαστε αντικειμενικοί, να μην προσανατεριστούμε κάποια συγκεκριμένη άποψη. Θέλουμε όμως να δούμε τις αντιδράσεις των πολιτών, του κοινού, ε, να έχετε κι εσείς μια αντικειμενική εικόνα για να μπορέσετε κι εσείς να προετοιμαστείτε κατάλληλα για την υιοθέτηση πολιτικών αποφάσεων. Τώρα για τη ε, τρίτη ερώτηση για τις προτεραιότητες. Έχετε απόλυτα δίκιο, όλοι το συζητάνε τώρα. Πρέπει να δούμε τι πρέπει μπορούμε να κάνουμε. Τα κράτη-μέλη δεν ε, συμφωνούν όλα πάντα και πολλές φορές ε, οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό είναι διαπραγματεύσεις για τις επιστροφές Γι' αυτό θα πρέπει τώρα, πιο συγκεκριμένα, λόγω και της ύφεση, ε, βλέποντας ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην ενέργεια και γενικότερα, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο γεγονός ότι η στρατηγική στόχη μας, ε, αυτό το οποίο θα πρέπει να πετύχουμε και εμείς και εσείς, είναι να προετοιμαστούν εγκαίρους τα στρατηγικά έγγραφα για την δημοσιονομική μεταρρύθμιση ερώτηση της κυρίας Μαγκίνες για την μεταρρύθ... μεταρρύθμιση ε, της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Την ερώτηση βέβαια την βλέπω με μια ιδιαίτερη έμφαση σε γεωργικά ζητήματα, αλλά έχει και γενικότερα χαρακτηριστικά που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τις γενικές παρατηρήσεις. Η δημόσια διαβούλευση που ξεκινήσαμε εμεί είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική γιατί ήταν η πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία που ε, ξεκίνησε τόσο ανοιχτά αυτή τη συζήτηση. Όποιο μπορούσε, όποιο ήθελε, μπόρεσε να συμμετάσχει σε αυτήν την διαβούλευση με κυβερνητικέ οργανώσει, κυβερνήσει, ε, ομάδε περισυλλογή, ε, οργανώσει πολιτών κτλ. Πολύ χρήσιμη λοιπόν και τώρα και στο μέλλον. Ταυτόχρονα όμω και εκφράζει βέβαια μεγάλο φάσμα ε, απόψεων και προοπτικών που δεν μπορούν να ε, περιοριστούν σε ένα μόνο μήνυμα. Γενικότερα βλέπουμε ότι υποστηρίζεται η προσέγγιση αυτή της μεταρρύθμισης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως μια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία για το κάθε ευρώ που δαπανάται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και προσφέρονται και κάποια κριτήρια για το πώς θα εξισορροπηθεί η σταθεροποίηση και η αποτελεσματικότητα του προπολογισμού. Πολλοί συμφωνούν ότι έχει ουσιαστικά εξελιχθεί αυτό ο προπολογισμό ε, σύν χρόνο. Λίγοι όμω είναι πολύ ικανοποιημένοι από την τρέχουσα δομή του προπολογισμού. Οι διαβουλεύσει λοιπόν μπορούν να δώσουν νέε προτεραιότητες ε, για τις προκλήσεις, κλιματολογική αλλαγή ιδιαίτερα και παγκόσμια ανταγωνιστικότητα ε, στο ύψιστο, στις πρώτες θέσεις του καταλόγου. Επίσης δημοσιονομικό σύστημα, τρόπος με τον οποίο παράγεται και εκτελείται ο οπισμός. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα βέβαια, τα αποτελέσματα τη διαβούλευση στην ιστοσελίδα μα. Και ιδιαίτερα για την ε, Γεωργία, από τη διαβούλευση βλέπουμε σχετικά ευρεία συνένεση ως προ την ανάγκη για αναθεώρηση τη κυρία γεωργικής πολιτική, αν και κάποιοι θεωρούν ότι θα πρέπει αυτή η μεταρρύθμιση να συνεχίσει αντίστοιχα με, ε, στην ίδια πορεία με το προηγούμενο check-up ενώ άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει πορεία η μεταρρύθμιση και θα πρέπει η κοινή πολιτική να επικεντρωθεί ή να ανταποκριθεί στις ανάγκες για ε, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια των προφήμων και σχετικές ε, ε, απαιτήσει κτλ. Διαφορετικές απόψεις υπάρχουν λοιπόν εδώ. Άρα η προσδοκίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση και με τους κύριες δαπάνες θα εξαρτηθούν και από τη διαβούλευση και από τις τεχνολογικές ε, αξιολογήσεις, επιστημονικές προτάσεις και ιδέες και θα είναι μέρο μέρος της πολιτικής απάντησης που θα δοθεί αργότερα μέσα στον χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε ένα στρατηγικό έγγραφο και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε σε συνεργασία και μαζί σας να ικανοποιήσουμε, να εκτελέσουμε σωστά αυτό το έργο. Ευχαριστώ, όλοι οι Πρόεδρος. Έχουμε τώρα την κυρία Μαγκίνες Φάρμ Παλέτης και ακούω την κυρία Μαγκίνες πρώτα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Επίτροπο τόσο για την απάντηση και για, τα σχόληση της, για την ε, ανταπόκριση της, ε, στην πρόταση της κυρίας Χάρκιν ως προς την ασφάλεια τροφίμων. Ένα μεγάλο πρόβλημα στην αγορά και θέλω ήθελα να επισημάνω και την έκθεση την οποία ψηφίσαμε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία, συντριπτική πλειοψηφία υπέρ τη ε, ΚΑΠ και τη ασφάλεια τροφίμων και ιδιαίτερα τα προβλήματα που έχουμε στο γαλακτοκομικό τομέα. Ότι χρειάζεται εδώ να επαληθευτεί η σχέση μα με την πραγματικότητα ω προ τι μεταρρυθμίσει αυτέ. Εδώ μιλούμε για τρόφιμα για τον Ευρωπαίο πολίτη, το εισόδημα αυτών που ζουν και διαχειρίζονται την ε, ε, υπεθρό μα. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε από κοινού. Κύριο Φάρμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία σύντομη ερώτηση προς την Επίτροπο. Ε, συμμετείχα στην εξαιρετική διάσκεψη που οργάνωσε η Κομισιό τον Δεκέμβριο για την δημοσιονομική μεταρρύθμιση και η Κομισιό ε, έκανε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για τις ε, προτινόμενες αλλαγές που θα υποβάλει. Όμως μετά την mid-term review ακούμε ότι δεν θα γίνουν αλλαγές και μετά τις ε, γερμανικές εκλογές και μετά τις ε, ε, εκλογές του για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Λοιπόν, πότε θα γίνουν οι τροπολογίες, πότε θα γίνουν οι προτάσεις της Κομισιόν για την αλλαγή, πριν ή μετά τις εκλογές. Κύριος Παλέσκης. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για, την τόσο, για τις τόσο συγκεκριμένες ε, απαντήσεις σας. Τα θέματα για την, ε, τις συζητήσεις για την δημοσιονομική μεταρρύθμιση ε, έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου και ήθελα να ρωτήσω πώς η οικονομική κρίση επηρεάζει τις συζητήσεις αυτές. Επίσης θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο θα ψάξτε να βρείτε κάποιες λύσεις για το πώς θα μπορούσατε δηλαδή να αποφύγετε τέτοιου είδου οικονομικέ κρίσει και αυτέ που ζούμε τώρα και στο μέλλον. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα ότι οποιαδήποτε απόφαση και αν πάρουμε στρατηγική απόφαση θα πρέπει να είναι πολιτική ε, και σίγουρη απόφαση. Πρέπει να είμαστε σίγουροι και για τον εαυτό μα. Δεν πρέπει να διακυβεύσουμε και να ε, διακρινεύσουμε οτιδήποτε από αυτά που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Απ' την άλλη πλευρά θα πρέπει να σα πω ότι ποτέ δεν μας είπαν ναι, ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα mid-term review για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Μας ζητήσαν να γίνει ένα, ένα κείμενο ε, ε, με μια πλήρη δημοσιονομική μεταρρύθμιση μέχρι το τέλος του 2009 και εμείς θα αποφασίσουμε πότε πολιτικά είναι πιο όριμη η συγκυρία για να υποβάλουμε το κείμενο αυτό, πότε θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική και υπεύθυνη απάντηση. Εγώ θα ήθελα να υποβληθεί το κείμενο αυτό εγκαίρως και γρήγορα την άνοιξη. Όμως δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι έχουμε πολλά πράγματα, τις εκλογές, την επικύρωση, την διαδικασία επικύρωσης της συνθήκης της Λισαβόνας και θα πρέπει ε, να μια καλή πρόταση να μην ε, την χαλάσουμε αν θέλετε ε, προβάλλοντας ταυτόχρονα και άλλα γεγονότα. Ας αποφασίσει ο κύριος Μπαρόζο. Τώρα, ήθελα να πω ότι η ερώτησή σας κύριε Πολέσκη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα ευρεία, πολύ ευρύτερη και από τα όσα μπορεί να προσφέρει ο κοινοτικός προϋπολογισμός η, παρούσα κρίση είναι τέτοια που κανένας ε, προϋπολογισμός και κανένα κράτος δεν θα μπορούσε να απαντήσει. Το πρόβλημα της κρίσης δεν προήλθε... Ε, τα προβλήματα που προκάλεσαν την κρίση δεν αφορούσαν ε, ε, τους προϋπολογισμούς ή τα, τα εισοδήματα, το ΑΕΠ κτλ. κτλ. Αφορούσε την ατέλεια ε, κάποιων μηχανισμών, επίβλεψης των ε, μηχανισμών. Και θα πρέπει να για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας περισσότερο σε μέτρα επίβλεψης και ελέγχου και μακροοικονομικά μέτρα και όχι τέλος πάντων στα ποσά αυτά καθεαυτά τα οποία θα βοηθούσαν για την καταπολέμηση της κρίσης. Υπάρχει το Ταμείο ε, παγκοσμιοποίηση, ή τέλος πάντων υπάρχουν κάποιες δυνατότητε που ε, δεν βοηθάνε άμεσα. Επομένως, ε, ναι, μεν τα σχέδια αποκατάστασης ε, αφορούν τη χρηματοδότηση κάποιων στρατηγικών μέτρων για, τα, για την ισοτομία της ενέργειας σε κάποιες υποδομές με, και έχει μια πρικοδότηση 5 δισεκατομμυρίων ευρώ τα κράτη-μέλη όμως δεν θέλουν να συζητήσουν τα project αυτά λόγω ακριβώς της κρίσης. Και η κρίση μας απέδειξε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρηματοδοτήσουμε και να επενδύουμε σε ε, ε, σχέδια υποδομών. Η κρίση νομίζω ότι αποτελεί ένα μάθημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μάθημα αυτό μας αποδεικνύει ότι θα πρέπει να, χρησιμοποιη... να δαπανούμε τα... τον προπολογισμό μας με έναν πολύ προσεκτικό και συγκεκριμένο τρόπο, διότι είναι μικρός ο προπολογισμό και δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα. Η παρούσα οικονομική κρίση και ύφαση θα πρέπει να βοηθήσει ε, τους πολιτικούς να ε, εστιάσουν περισσότερο προσοχή στις επενδύσεις. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε τώρα στην ερώτηση προς τον κύριο Ζακ Μπαγό. Έχουμε 16 ερωτήσεις. Προφανώς δεν θα α, ε, ακουστούν ε, και οι 16 ερωτήσεις, οι τρεις πρώτες που ήρθαν. Ε, ερώτηση του κυρίου Νιχτένε για την ε, εγκληματικότητα online. Ευχαριστώ πολύ κύριε, Πρόεδρε. Θα απαντήσω στο ερώτημα που ετέθη, ερώτημα του κυρίου Νέχτη για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Εμείς καταπολεμούμε εδώ και χρόνια το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Το κάνουμε σε στενή συνεργασία με, την, με τα κράτη-μέλη και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν συμμετέχει με τέσσερις τρόπους στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον χώρο. Καταρχάς προωθώντας ε, τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, διευκολύνοντας ε, τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αναπτύσσοντας ε, διάφορα νομικά εργαλεία και ξεκινώντας μια συνεργασία με τα, κράτη, με τα τρίτα κράτη, με τις τρίτες χώρε Η Κομισιό, και μάλλον στην ανακοίνωσή της του 2007, με τίτλο προς μια γενική πολιτική με στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Ε, μπορέσαμε να προωθήσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο είτε, διμερός, με διμερή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, είτε μέσω της Europol. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουν μόνιμα σημεία επαφής ε, μέσω των οποίων τα άλλα κράτη-μέλη μπορούν να τους, να τους ζητήσουν βοήθεια ή πληροφορίες. Η Κομισιό επίσης έχει συμμετάσχει στην ε, σύνταξη συμπερασμάτων του Κοινοβουλίου ε, που υιοθετήθηκε πέρυσι τον Νοέμβριο για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Η στρατηγική αυτή προτείνει μια ολόκληρη σειρά μέτρων που έχουν σαν στόχο να ε, ενισχύσουν τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τα, και την καταπολέμηση εγκλημάτων όπως η τρομοκρατία, παιδεραστία και απάτες, καταπολέμηση των απατών. Ε, δημιουργείται μια πλατφόρμα πληροφοριών στο ίντερνετ που θα πρέπει να ε, να ομαδοποιηθούν τα εγκλήματα αυτά από την Europol. Επίσης, η η Κομισιόν ε, προωθεί μια συνεργασία ανάμεσα στις κατασταλτικές αρχές και ε, τον ιδιωτικό τομέα για την καταπολέμηση του εγκλήματος των κυβερνοχώρων. Το Συμβούλιο Τζάι της 8 ε, Δεκεμβρίου του 2008 ε, κατέληξε σε συστάσεις για την ε, συνεργασία ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την καταπολέμηση του κλίματος στον κυβερνοχώρο. Η Κομισιόν θέλει να εφαρμόσει, μια, ε, να δημιουργήσει μια οικονομική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της χρήσης των, της παιδεραστίας για τις διαφημιστικούς λόγους. Θέλουμε να ε, απαγορευτεί η δημοσίευση φωτογραφιών ε, παιδοπορνογραφικού περιεχομένου στο ίντερνετ. Η Κομισιόν συμμετείχε ε, σημαντικά στην δημιουργία μιας ενός νομοθετικού πλαισίου που, δημιουργούν ελάχιστες προδιαγραφές για την εναρμόνιση της νομοθεσίας, παραδείγματος χάρη απόφαση πλαίσιο ε, του 2005 για, την, ε, για τις επιθέσεις των συστημάτων ενημέρωσης και πληροφόρησης, ε, απόφαση πλαίσιο του 2004 για το GIE, για την καταπολέμηση της παιδοπορνογραφίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Η Κομισιόν εξετάζει τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε όλες, όλα αυτά τα εργαλεία. Και καταλήγω λέγοντας ότι το ίντερνετ είναι ένα, ε, ε, σύστημα που μας επιτρέπει ε, να διακινηθούν πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί από μόνη της να ρυθμίσει το ίντερνετ. Γι' αυτό η Κομισιόν θα ήθελε να προωθήσει μια διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτό και θα οργανώσουμε φέτος μια, μια συνάντηση με διεθνείς φορείς και με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να συντονιστούν οι δράσεις όλων αυτών των διεθνών, οργασιών, των, των διεθνών οργανισμών αλλά και των υπευθύνων κοινοτικών φορέων. Αυτά μπορώ να απαντήσω στον κύριο Νέχταν. Και πάντα για να προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο θα ενώσω, ενωπίσω τις συμπληματικές ε, ερωτήσεις ο Νάχταν και τη Τσάου. Παρακαλώ κύριο Νάχταν. Και μετά το... Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την απάντησή του και θα ήθελα να καταθέσω μια συμπληρωματική ερώτηση. Κύριε Επίτροπε, για τον εκφοβισμό, το λεγόμενο bullying μέσω του κυβερνοχώρου. Ιδιαίτερα θύματα του είναι τα παιδιά και οι νέοι που χρησιμοποιούν ε, το Flickr και το Facebook. Ενισχύονται όμω τέτοια φαινόμενα, εντείνονται τέτοια φαινόμενα αυτό ο εκφοβισμό μα του κυβερνό και ρωτώ τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει περισσότερη προσοχή, ε, περισσότερη σοβαρότητα στην αντιμετώπιση αυτού του ε, εκφοβισμού. Κύριε Τιτσάο και μετά του κύριο Στόβερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Στο επόμενο ερώτημα λοιπόν θα ήθελα να μου απαντήσει ο Επίτροπος τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή ώστε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εγκληματικότητα μέσω του κυβερνοχώρου τι δράση σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εισαγάγει για να βελτιώσει την ε, ε, αντιμετώπιση της εγκληματικότητας μέσα στον κυβερνό χώρο. Και επίσης για την ηλεκτρονική υπογραφή θα ήθελα να μου πείτε αν σκοπεύετε να προχωρήσετε στην γενικευσή της. Ο κύριος Ντόβερ παρακαλώ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ευχαριστήσή μου προς τον σε ευχαριστήσουμε μάλλον προς τον Επίτροπο για την απάντηση που μας δίνει, αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα να μιλήσουμε και τον κόσμο συγκεκριμένα. Εγώ είμαι υπέρ βέβαια της πάταξης του κυβερνοεγκλήματος. Ωστόσο δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι εταιρείε του ίντερνετ δεν θα πρέπει, όπως άλλωστε και η αστυνομία και οι λοιπές αρχές, να επιβάλλουν υπερβολικά ε, αυστηρίες συνθήκες χρήσης του ίντερνετ που είναι και μέσω αναψυχής. Ο Επίτροπος βεβαίως και έχετε δίκαιο Απαντώ αμέσως στην ερώτηση σχετική με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πάταξη του κυβερνού εγκλήματος. Βεβαίως πρέπει να, έχουμε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτός ο αγώνας κατά της, του κυβερνού εγκλήματος να γίνει με κάθε σεβασμό ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και για να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, στο δε πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα συμπληρώσω πολιετε προγραμμα πρόγραμμα 2010-2014 έχουμε ενσωματώσει όλο αυτό το κεφάλαιο, ολόκληρο ένα κεφάλαιο για την ε, πάταξη του κυβερνοεγκλήματος και όπως είπα και νωρίτερα και προς τον κύριο Νάκταν, υπάρχει σαφής βούληση για ένα κέντρο για ένα παρατηρητήριο υπό την Europol που θα μας επιτρέπει να παρακολουθούμε καλύτερα και να συντονίζουμε την εποπτεία των εθνικών ε, θεσμών που, στόχο έχουν, ε, που καθήκον έχουν την εποπτεία και παρακολούθηση των ύποπτων. σελίδων ή χώρο ιδιαίτερα όταν θύματα είναι παιδιά ή γενικά οι πληθυσμοί ευάλωτοι βάλει ομάδες πολιτών. Όπως είπατε και εσείς υπάρχουν ε, διάφορα sites ε, στα οποία κινδυνεύουν ε, οι νέοι από επιθετική συμπεριφορά και εκφοβισμό. Αυτές είναι οι απαντήσεις που μπορώ να δώσω. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να πω ότι έχουμε δράσεις να αναπτύξουμε με πιο αποφασιστικό ακόμη τρόπο από ότι στο παρελθόν, αφού γνωρίζουμε και καλύτερα τους κινδύνους του διαδικτύου. Αυτά έχω να σας δώσω ως απαντήσεις και πιστεύω ότι και η οικονομική αλληλεγγύη, μάλλον συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ε, στον οικονομικό εμπορικό χώρο της διάθεσης ε, εικόνων παιδικής πορνογραφίας μέσω του διαδικτύου θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ. Εάν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση μέσα από, μέσα από την Επιτροπολογία, μπορούμε να, να ξεκινήσουμε τη λειτουργία αυτού του συστήματος από το Φεβρουάριο του 2009 και ελπίζω το Κοινοβούλιο να μας υποστηρίξει. Και τώρα, λέει η Πρόεδρος, έχουμε την ερώτηση του κυρίου Έλουαρτ. Τρομοκρατικές απειλές, απειλές τρομοκρατικών επιθέσεων. Κύριε Επίτροπε. Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας απαντώ ως εξής, αγαπητέ κύριε. Για να μπορεί κανείς να καταπολεμήσει η τρομοκρατία και το σοβαρό έγκλημα γενικότερα είναι το ότι θα πρέπει να υπάρχουν την κατάλληλο χρόνο οι πληροφορίες που χρειάζονται, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι τεράστια πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και προσπαθήσαμε να προωθήσουμε την διευκόλυνση της και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αστυνομιών και των μελών. Η δε απόφαση πλαίσιο της 18ης 12 του 2006 ε, η λεγόμενη σουηδική απόφαση αφορά το ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει μέχρι το 2008 να έχουν, δηλαδή που να έχουν ένα κοινό πλαίσιο τόσο να υπάρχει ταχύ ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και κρατομερών για αυτό το σκοπό. Και αυτή η απόφαση πλαίσιο απαιτεί οι αστυνομίε των κρατών οι οποίε δέχονται με ένα σχετικό αίτημα, θα πρέπει να το διεκπεραιώνουν χρησιμοποιώντα κάποια κριτήρια τα οποία θα πρέπει να είναι σύντονα με αυτά τα οποία ισχύουν και για τις ε, εθνικές ε, έρευνες και ανακρίσεις. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο είναι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της 23 έκτου του 2008. Προβλέπεται λεπτομερής ενδελεχής μηχανισμός για την ανταλλαγή ε, συγκεκριμένης κατηγορίας δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων του DNA ε, σχετικά με τους αριθμούς κυκλοφορία των αυτοκινήτων, όλε αυτές τι πληροφορίες, ώστε να είναι δυνατόν να διεκπεριωθούν οι έρευνε για εγκλήματα. Και δυνάμει αυτή τη αποφάση του Συμβουλίου. Τις αποφάσεις Ντεπρέμ, τα κράτη-μέλη έχουν περιορισμένη προσβασιμότητα στα δεδομένα DNA και στα ε, δακτυλικά αποτυπώματα ώστε να ε, δουν κατά πόσο υπάρχει ταύτιση. Και έτσι με αυτή την απόφαση του Συμβουλίου να δούμε έχουμε αποτελεσματική ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών για το DNA και για τα αποτυπώματα η Europol. Επίσης έχει κρίσιμο ρόλο σε αυτή την υπόθεση το σύστημα πληροφοριών της Europol, το SIE, επιτρέπει στα κράτη-μέλη να καθορίσουν κατά πόσον οι διοκτικές αρχές έχουν τις ε, απαραίτητες πληροφορίες σε επίπεδο επιχειρησιακό. Όμως, βέβαια, για να μπορεί να κάνει τη δουλειά της Europol θα πρέπει τα κράτη-μέλη να τροφοδοτούν αυτό το σύστημα πληροφόρησης με τρόπο αποτελεσματικό. Βεβαίως. Και θα πρέπει να δούμε πως κάποια στιγμή θα τεθούν σε ισχύ νέες διατάξεις για να υπάρχει ανταλλαγή πληροφόριων σε αυτό το πενταετές πρόγραμμα το οποίο θα διαδεχθεί το πρόγραμμα της Χάγης το οποίο θα πρέπει να υπάρχει εγγύησης για κάποια συντονισμένη προσέγγιση συνεκτική όσον αφορά τις ε, πληροφορίες. Επίσης θα πρέπει σε αυτό το πενταετές ε, πρόγραμμα να περιληφθεί και κάποια ενωσιακή στατική ανταλλαγή πληροφοριών βεβαίω. Όμω, ανταλλαγή πληροφοριών σημαίνει και ταυτόχρονα προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η δε στρατηγική θα πρέπει να επιτρέπει μια σφαιρική προσέγγιση του θέματος, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε και στις αστυνομικέ ανάγκες και που θα πρέπει να είναι διαλειτουργική όσον αφορά τα διαφορετικά συστήματα, όσον αφορά ε, το τεχνολογικό επίπεδο. Ναι, αυτά τα στοιχεία μπορώ να σας απαντήσω. Και κύριε Aylward. Θα μαδοποιήσω τις ερωτήσεις επομένως. Κύριος Hailward, κύριε Ντόιλ, Κύριε κύριος Ζούμπικε, κύριος Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την απάντησή του. Μία πολύ σύντομη συμπληρωματική ερώτηση. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ναι, την κατάσχεση των ε, ε, στοιχείων του ενεργητικού, των, ε, των περιουσιακών στοιχείων των τρομοκρατών στην Ευρώπη. Διότι θεωρούμε ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Ντόιλ, ευχαριστώ πολύ ε, θα ήθελα η Κομισιό να μας πει αν εξασφαλίζει τη συνεργασία και των 27 κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και αν όχι ποιες είναι οι χώρες που ακολουθούν διαφορετική γραμμή και η Ιρλανδική κυβέρνηση ζήτησε ε, ε, ένα opt-out στον τομέα αυτό, ο κύριος Ρούμπικ. Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, Υπάρχει κάποια έννοια διασφάλισης, ασφάλειας ως προς τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ο Επίτροπος. Ως προς την ε, κατάσχεση αγαθών που αποτελούν παράνομο προϊόν, προϊόν εγκλήματος από αυτά τα, στο μελετούμε εμβριθώς τα θέματα αυτά. Ο Ζων Μπρίκερ, ιδιαίτερος έχει επιληφθεί τις εποπτείας του προγράμματος SWIFT της ε, παρακολούθησης και ανείχνευσης της τρομοκρατίας. Σύντομα θα έχω τα πορίσματά του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την χρηματοδότηση από την αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος και βέβαια ο δικαστής Μπρούχερ χρησιμοποιεί, αξιοποιεί στο μέγιστο τα ποσά που του διατίθενται. Όπως είπα, πρόκειται για την ε, κατάσχεση αγαθών που αποτελούν ε, ατόμων που έχουν ε, εξασφαλίσει κέρδος από εγκληματικές πράξεις. Με η λειτουργία της Europol θα πρέπει να σας πω θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική αν μας δίθεταν και τα κράτη-μέλη πιο γενναιόδωρα και με τρόπο πιο διαφανή τις πληροφορίες που χρειάζονται. Ιδιαίτερα λοιπόν με απασχολεί το πώς θα δημιουργήσουμε αυτή την έννοια της εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών που επιλαμβάνουν των θεμάτων αυτών μεταξύ των κρατών μελών για να έχουμε πιο αποτελεσματική δράση. Για ρήτρα εξαίρεση δεν μπορώ να μιλήσω, δεν έχω ακούσει τίποτα στον τομέα αυτών. Μάλλον ε, απάντησα εντωμεταξύ στι ερωτήσεις σας. Τώρα για την πυρηνική απειλή, για απειλέ ε, κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων. Έχουμε φροντίσει για ένα κείμενο ε, που καλύπτει τις κρίσιμου χαρακτήρα υποδομές, όπως ονομάζονται, με τι οποίες εγκαταλέγονται και οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει ένα κείμενο που επιτρέπει καλύτερη εποπτεία, παρακολούθηση, έλεγχο των ε, ε, κρίσιμων ε, υποδομών. Τελευταία ερώτηση για τον κύριο Μπαρό τώρα, από τον κύριο Φράνσα για τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ. Λοιπόν, απαντώ στον κύριο Φράνσα, Φράνκα η σφαιρική προσέγγιση προς την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει να δώσει μια γενική απάντηση στην πρόκληση που δημιουργεί το μεταναστευτικό ρεύμα στην Ένωση. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τον διάλογο και τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, αυτή είναι η προσέγγισή μας, σε, για όλες τις πτυχές της μετανάστευσης, έτσι ώστε να υπάρξει μια συνεργασία αποτελεσματική για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης για να δώσουμε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο σε αυτή την σφαιρική προσέγγιση στον τομέα της μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ε, συνεργασίες με τις τρίτες χώρες για τη μετανάστευση και το άσυλο. Παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα ΕΝΑΣΑ, το οποίο χρηματοδότησε πάνω από 100 project στην ε, περίοδο 2004-2006 ή επίσης το πρόγραμμα ε, για τη μετανάστευση και το άσυλο που ακολούθησε ήταν 205 ε, εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2005-2010. Ανάμεσα σε όλες αυτές ε, τις προτεραιότητες ε, που υιοθετούνται μέσα στα πλαίσια ετήσιων εξετάσεων, πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες προτείνονται και εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Με βάση το πρόγραμμα ΑΕΝΑΣ, η Κομισιό χρηματοδοτεί ένα project της Ισπανίας και του Μαρόκου για τον έλεγχο της εποχιακής μετανάστευσης ανάμεσα στις επαρχίες Μπεν Σλιμάνα και της Ουέλβα στην Ισπανία. Στο Μαρόκο και στην Ισπανία αντίστοιχα. Το ίδιο το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει και τη συνεργασία ανάμεσα στην Ισπανία και στην Κολομβία για να αναπτύξουμε μια κυκλική μετανάστευση. Επίσης, χρηματοδοτήσαμε την προσωρινή επιστροφή υπηκών του πράσινου ακροτηρίου που είχαν ε, προσόντα ε, και που βρίσκονταν στην Πορτογαλία και επέστρεψαν στο ΚΑΠ Βέρντε, στο πράσινο ακροτήριο, έτσι ώστε να εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν δυνάμει υποψήφιους μετανάστες. Πέραν αυτών των παρεμβάσεων, Έχουμε και οικονομικά, γεωγραφικά μέσα, παραδείγματος το μέτρο ε, γυτνίασης ε, που ευνοεί αυτή την σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης. Παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε πρόσφατα την εφαρμογή και τη δημιουργία ενός κέντρου ε, πληροφόρησης για τη μετανάστευση στο Μαλί. Είναι ένα project στο στο οποίο συμμετέχουν και πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μέσα στα πλαίσια της ε, σφαιρικής προσέγγισης, η Κομισιόν πρότεινε νέα εργαλεία για να ευνοήσουμε τη συνεργασία με τρίτες χώρες και για να αναπτύξουμε κάποιες ε, πιο στενές συνεργασίες ανάμεσα στην, στις, στα κράτη-μέλη και στην Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνεργασίες για την κινητικότητα που είναι ένα νέο εργαλείο ε, το οποίο εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πιλωτικά σε μια πρώτη φάση και αυτές ε, οι συνεργασίες για την κινητικότητα επιτρέπουν ε, την ανάπτυξη ενός διαλόγου, μια συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, της ανάπτυξης, της πρόληψης και της μείωσης της παράνομης μετανάστευσης. Έχουμε υπογράψει επομένως ε, πρώτες συνεργασίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πράσινο Ακροτήριο και την Δημοκρατία της Μολδαβίας. Μέσα στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών Έχουμε διατυπώσει συγκεκριμένες προσφορές συνεργασίας. Παραδείγματο χάρη, στον τομέα τη συνεργασία με το Πράσινο Ακροτήριο, η Πορτογαλία πρότεινε την υπογραφή ενό νέου πρωτοκόλου ε, που παρατείνει ένα ισχύον πρωτόκολλο για την προσωρινή μετανάστευση ε, εργατών από το Πράσινο Ακροτήριο που θα έρθουν να εργαστούν στην Πορτογαλία. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Υπάρχει το, ο, ο μεταναστευτικό απολογισμό που αναλύει την μεταναστευτική κατάσταση κάποιες δεδομένε χώρας. Υπάρχουν πλατφόρμες συνεργασίας επίσης που ε, επιτρέπουν τη συγκέντρωση ε, των ε, ενδιαφερομένων σε μια χώρα όπως επίσης και των σημαντικότερων χρηματοδοτών. Έχουμε δημιουργήσει μια τέτοια πλατφόρμα συνεργασίας στην Αιθιοπία με πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου ε, προβλέπουμε να δημιουργηθεί μια άλλη πλατφόρμα στην Νότια Αφρική. Υπάρχει το Ταμείο Ένταξης και το Ταμείο Επιστροφής που βοηθάνε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να δημιουργήσουν στα στις τρίτες χώρες ε, μέτρα πριν από την αναχώρηση έτσι ώστε να, βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι δυνατότητες ένταξης του εργαζομένου που θα μεταναστεύσει σε μια χώρα μας ή επίσης που θα διευκολύνουν την επιστροφή του ενδιαφερομένου. Αυτά, ε, κύριε Βουλευτά, είναι ορισμένα παραδείγματα. Όμως να σας πω ότι είμαι απόλυτα πεπισμένος για την ανάγκη για την Ευρώπη να διαχειριστεί τα μεταναστευτικά ρεύματα με αυτή την ε, γενική προσέγγιση που συνδέει τα θέματα ανάπτυξης και μετανάστευσης και που επιτρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη ε, διαχείριση της μετανάστευσης. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος τον οποίο θα πρέπει να έχουμε και ε, θα δημιουργήσει ένα παράδειγμα για όλους ομαδοποιώ τις ερωτήσεις ο κύριος Φράνσα και μετά ο κύριος Πέρτα. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Μπαρό, συμφωνώ με τα όσα μας εξηγήσατε, αλλά επίσης συμφωνώ με το ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και οίκιστα ικανοποιημένοι από όλα αυτά τα μέτρα. Μια που η λάθρομετανάστευση συνεχίζει να σοβεί στην Ευρώπη. Έχουμε αυτό το δουλεμπόριο το οποίο επίσης συνεχίζεται και έχουμε τόσες περιοχές όπως στην Μεσόγειο, στην Ιταλία και στη Γαλλία όπου υπάρχει πολύ έντονο αυτό το πρόβλημα. Έχουμε διάφορα μέτρα που έχουν ληφθεί, έχουμε και διμερεί μέτρα, αλλά πολλά κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν. Τι λέτε, να δείτε πώς θα συνεχίσει το έργο του Ευρωπαϊκής Πρόεδρος. Έχουμε πάρα πάρα πολύ καθυστερήσει. Έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η ερώτηση αναφέρεται στον ανθρωπιστικό στοιχείο αυτή τη ε, πολιτική μετανάστευση και την εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί είχαμε ε, πρόσφατα την έκδοση κάποιο παρά το ότι ε, υπήρχε απειλή γενετήσιου ακροτηριασμού των θυγατέρων του. Τέλος πάντων, τι γίνεται αυτό δεν είναι πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφού είναι έτσι τα πράγματα δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξωθεί στα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν κατάλληλη νομοθεσία με αυτή την κοινή θέση. Ο κύριος Επίτροπος, να σας ε, απαντήσω, ο κύριε Φράγκα, ότι θα κάνω ό,τι μπορώ, ούτως ώστε να έχουμε μια συνολική προσέγγιση μέσω εταιρικής σχέσης για την κινητικότητα από τη μία να είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη τρίτε χώρε για μια τέτοια συμφωνία. Βεβαίω κάποια κράτη-μέλη κατάφεραν να συνάψουν τέτοιε διμερεί συμφωνίε. Αλλά αυτό θα πρέπει να ισχύσει για όλου στην Ευρώπη. Μια που, εάν δεν έχουμε καλή οργάνωση τη ε, νόμιμη μετανάστευση, ε, υπάρχει μεγάλη επιλογή μετανάστευση. Άκουσα ότι είπατε κύριε Βουλευτά, ε, αυτό το πράγμα το οποίο αναφέρατε καταδεικνύει ότι η πολιτική του επαναπατρισμού θα πρέπει να γίνεται κάνοντας κάποιες λεπτές διακρίσεις. Δεν είναι δυνατόν να στέλνουμε τον κόσμο σε κάποια κράτη, τρίτα, τα, όταν απειλούνται, απειλείται η ακυριότητά τους, η ζωή τους, θα πρέπει επομένω να επιδείξουμε πιο δύναμη διάκρισης. Γιατί έχουμε εδώ πέρα <clears throat> Ε, αυτό το, το, το, το νομοθέτημα ε, θα πρέπει βέβαια αυτό το νομοθέτημα ως οδηγία να το αναδεχθούν σωστά τα κρατη αλλά έτσι θεωρούμε ότι θα βελτιωθεί η πολιτική του επαναπατρισμού. Θα παρακολουθήσουμε εξελίξεις με προσοχή 38 με 50 είναι ερωτήσεις οι οποίες εγγράφως θα απαντηθούν. Πάμε τώρα η ερώτηση που αφορά τον Επίτροπο κ. Μακρύβη. Η πρώτη ερώτηση. Είναι η ερώτηση κυρίου Αγγελάκα και αφορά το άνοιγμα στην αγορά των κλειστών ευαγγελμάτων. Αν θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η Κομισιό δεν έχει σαν στόχο να είναι το άντεγμα κλειστών επαγγελμάτων. Μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής ε, πολιτικής υπάρχει το άνομο συμφέρον των κρατών μελών να ε, διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελμάτων. Θα πρέπει να δούμε ποιος, και είναι στις συνέπειες και στην ευρωπαϊκή ε, οικονομία. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε την, ε, τις εθνικές νομοθεσίες και να δούμε κατά πόσον υπάρχουν αυθαίρετοι περιορισμοί στην πρόσβαση σε κάποια απεγγέλματα. Επίσης υπάρχει και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ούτως ή άλλως θα πρέπει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν συγκεκριμένη ημερομηνία, μια έκθεση στην ε, Κομισιό για το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, ε, δηλαδή της ε, αξιολόγησης των εθνικών νομοθεσιών και την, της εφαρμογής αυθαίρετων περιορισμών για την πρόσβαση σε κάποια επαγγέλματα και με τον τρόπο αυτό ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιου είδους αυθαίρετες, περιορισμοί και ενδεχόμενα θα πρέπει να συζητήσουμε και τις απαραίτητες αλλαγές που απαιτούνται στην νομοθεσία κάποιων κρατών μελών. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2010 η Κομισιόν θα υποβάλει μια σύνοψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, στην, και στο Συμβούλιο για την αποτελέσματα αυτής της κοινή αξιολόγησης που θα γίνουν και τότε θα συζητήσουμε και το περιεχόμενο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λειτουργεί η εσωτερική αγορά και έχουν, εφόσον υπάρχουν εθνικοί κανόνες που εφαρμόζουν μέτρα διακριτικής μεταχείρισης, ξεκινάνε, ξεκινάει και η διαδικασία έρευνας. Η Κομισιόν στον τομέα του ανταγωνισμού προσπαθεί να αναθεωρηθούν ε, οι επαγγελματικοί κανόνες που ισχύουν στα κράτη-μέλη. Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού καλούνται υπό το φως των κανόνων ανταγωνισμού να εξετάσουν την κατάσταση και ελπίζουμε ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Θα ακούσουμε τι ερωτήσει τώρα πάλι ενωποιημένο ο κύριο Αγγελάκα, ο κύριο Ρούβιχ και η κυρία Ντόιλ. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που θέλει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή είναι η δημιουργία μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς και ελεύθερης διακίνησης επαγγελμάτων. Από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που εγώ τα αποκαλώ κλειστά, τα οποία, για τα οποία την άσκηση των οποίων έχουν καταβληθεί ποσά και αναφέρομαι σε άδειε ταξί που σε πολλέ χώρε κράτη μέλη της Ευρώπη είναι κοστολογημένες όπως επίσης το φαρμακευτικό επάγγελμα όπου αυτό ασκείται με πληθυσμιακά και αποστασιακά μέτρα. θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις του επιτρόπου. ότι τοπικού χαρακτήρα και περιφερειακές προδιαγραφές μπορεί να αποτελούν βασικό όρο βάσει το οποίο μπορεί να ασκηθεί το επάγγελμα. Κύριε Ντόιλ. Ευχαριστώ δεν ξέρω αν οι tour operators και οι bookmakers, αυτοί που, που δουλεύουν σε γραφεία στοιχημάτων, υπάγονται στην ίδια κατηγορία, αλλά πάντως για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την παροχή των υπηρεσιών στην ιστορική αγορά, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τους συστήσουμε και αυτούς. Υπάρχουν ε, τέτοιου είδου πληροφορίε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων με τη σχετική οδηγία και την έννοια τη αμοιβαία ε, αποδοχή των ε, δεξιοτήτων έχει προχωρήσει καθόλου από το ένα κράτος στο άλλο. Ο Επίτροπος. Εδώ έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα. Πρώτον, το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία των υπηρεσιών και δεύτερον, η υπηρεσία περί επαγγελματικών προσόντων. Η οδηγία περί υπηρεσιών ασχολείται γενικά με τις υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ λίγες περιορισμένες εξαιρέσεις. Ο κύριος Αγγελάκα, μίλησε για τις ε, για του φαρμακοποιού. Θα γνωρίζετε ασφαλώ ότι υπάρχουν κάποιε διαδικασίε σε παραβιάση ε, κατά ορισμένων κρατών μελών για την παραβίαση των διατάξεων. Και κάθε κράτο μέρο έχει την υποχρέωση υπό την οδηγία περί υπηρεσιών να προσαρμόσει τις διατάξεις και η νομοθεσία του πριν από το Δεκέμβριο του 2000 φέτος για να γίνει στη συνέχεια η αμοιβαία αξιολόγηση του κατά πόσο αναλογικά είναι σκόπματα όσα έχουν προταθεί. Ε, για δε κυρία Ντόιλ. Στα θέματα της παραβίασης των κανόνων περί χαρτοπεξίας, ε, στοιχημάτων κτλ. Έχουμε νομοθεσία, νομολογία συγγνώμη, ως προς την υπηρεσία αυτή που αναγνωρίζεται ως υπηρεσία δηλαδή, το στοίχημα, η το κτλ. Και θα πρέπει να επαχθεί και αυτή στην οδηγία περί υπηρεσιών και άρα αντίστοιχα θα πρέπει να κινηθούν διαδικασίες παραβιάσεις κατά των κρατών μελών εφόσον υπάρχουν παραβιάσεις των διτάξεων της οδηγίας η Πρόεδρος. Καλώς προχωρούμε στην ερώτηση του κυρίου Παπαστάμκου. Οργανισμοί επιφορτισμένοι με την πιστοληπτική ικανότητα, αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Παρακαλώ τον Επίτροπο να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγες δραστηριότητες τέτοιων οργανισμών τα τελευταία χρόνια και ύστερα από το ψήσιμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου του 2004 εξετάζει με πολύ μεγάλη προσοχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον ε, νομοθεσία για την παρακολούθηση των ε, ε, οίκων αξιολόγηση πιστολιστικής ικανότητας. Είχαμε μια πρόταση το Μάρτιο 2005 και στο 2006 το Μάρτιο υιοθέτησε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία καταλήξει το συμπέρασμα ότι, ορισμένες, ότι διάφορες μάλλον οδηγίες περί υπηρεσιών καλύπτουν και τους σχετικούς οίκους αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και υπάρχει βέβαια και κώδικα συμπεριφοράς που μπορούν να δώσουν α, ικανοποιητικές πιστεύουμε απαντήσεις στις όποιες ανησυχίες ως προς τη λειτουργία αυτών των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Βέβαια παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της, ε, την κατάσταση και τις εξελίξεις και ενημερώνει τακτικά, ετησίως δηλαδή. Από την άλλη, από την ανακοίνωση λέγεται, σημειώνεται ότι μπορεί να εξετάσει αν υπάρξει πρόβλημα τήρησης των σχετικών διατάξεων ή αν προκύψουν νέες συνθήκες θα μπορούσε σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων, ε, μη ομαλής λειτουργία τη αγορά, ε, να εξετάσει και τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται τέτοιου είδου οίκοι ανά τον κόσμο σε διαφορετικέ χώρε δηλαδή. Ύστερα από το μεγάλο πρόβλημα της κρίσης εμπιστοσύνης ως προς τις φωτοπιστικές αγορές το 2007 και μετά βλέπουμε ότι αυτή η αξιολόγηση βρίσκονται κοντά στα προβλήματα που προέκυψαν με τις αγορές των subprimes. Έχουν δηλαδή συνάφεια με αυτά τα προβλήματα και ήταν μη ικανοποιητικό ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν συγκρούς συμφερόντων αυτή η αξιολόγηση αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Οι αδιαφάνειες προς τη δραστηριότητά τους ε, αποδεικνύουν ότι δεν ήταν ικανοποιητική η επιχειρηματική διαχείριση αυτών των οίκων και πρέπει να ενισχυθεί η παρακολούθηση της λειτουργίας τους. Γι' αυτό τον λόγο, τον Ιούνιο του 2008 ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα αναλάβει κανονιστική δράση. Το Δεκέμβριο του 2008 με τους αδέλφους υιοθετήσαμε πρόταση που ρυθμίζει την δραστηριότητα αυτών των οίκων αξιολόγηση με συμφωνία βέβαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θα δω τώρα, θα ακούσω μάλλον τώρα και τους δύο ε, συντάκτης, τον κύριο Παστάπ και τον κύριο Ρερ. Επίτροπε, εσείς ο ίδιος το 2006, απαντώντας σε σχετική μου ερώτηση, μου είπατε επιλέξει ότι σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, η Επιτροπή, δηλαδή η Κομισιόν, δεν υποβάλλει νέες νομοθετικές προτάσεις στον τομέα των οίκων διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας. επισυνέβη η μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση και ήρθατε τώρα να μας πείτε ότι χρειάζεται αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. πράγματι χρειάζεται αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. το ερώτημά μου αναγνωρίζετε αμβλημένα ρυθμιστικά αντανακλαστικά της κομισιόν επί του θέματος αυτού. Monsieur Thank Σας ευχαριστώ, Λίγης Ράιν. Um, Έχουμε αυτές τις πρωτεύουσες επιτροπής για την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Κάτι το οποίο ε, ε, κάπως θα ωφελήσει τους αποταμιευτές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γιατί μπορεί να κάνει τούτος ώστε να βοηθήσει την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα στην πραγματική οικονομία και κυρίως όσον αφορά τον κλάδο των ΜΜΕ, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα, τώρα που λένε και περισσότερο πλήρως της ευρωπαϊκής οικονομίας, στα φαινόμενα της ύφεσης. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Για τον κύριο Παπαστάμκο. Έχουμε την στο το 2005 ε, στα πλαίσια της οποίας προβλέπεται αυτοί οι φορείς να ασκήσουν μία εποπτεία και το 2007 φτάσαμε στην κορύφωση της κρίσης με την αγορά των subprimes και είχαμε πει τότε για, αυτές τις, για αυτούς τους φορείς ότι δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι σε σχέση με το πώς επιτελούν τα καθήκοντά τους και θα γνωρίζει ο κ. ότι το Δεκέμβριο του 2007 και στη ΣΥΖΑ και στην ΕΣΜΕ είχα απευθυνθεί διεπιστολή μου σε σχέση με το θα πρέπει να διερευνήσουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα και ε, είχαμε πει ότι το να μείνουν τα πράγματα όσο έχουν τότε, αυτό το status quo το τότε είναι κάτι το απαράδειτο, δεν είναι καμία λύση, οπότε τελικά ε, το 2008 εκπονήσαμε αυτή την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρότασή μας την έχουμε υποβάλει αρμοδίω σε εσάς και στο Συμβούλιο των Υπουργών. Και στο παρελθόν, στα πλαίσια της αναθεώρησης των όσων διέπουν αυτούς τους οργανισμούς αξιολόγησης της στρατιωτικής ικανότητας, είπαμε ότι στη συγκυρία αυτή όπως είχε τα πράγματα δεν ήταν εντάξει. Δηλαδή άραξαν τώρα τα δεδομένα και άρα θα πρέπει να αλλάξει η λειτουργία αυτών των φορέων. Ο κ. Ράιν ερώτησε πέραν αυτών των μέτρων, των ρυθμιστικών, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους φορείς, για αυτούς τους οργανισμούς. Ρώτησε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχετε δίκιο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την οικονομία. θεωρούμε ότι η αλλαγή, οι αλλαγές που κάναμε στον ημεσονικό κανονισμό θα θωρακίσουν την ευρωπαϊκή οικονομία και θα άρουμε κάποια κενά που υπήρχαν σε αυτές τις ρυθμίσεις. Προσπαθούμε να έχουμε έναν συντονισμό στις προσπαθίες μας για να βοηθήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Έγινε κάποια προσπάθεια και στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου Βέβαια και τα κρατη θα πρέπει κάτι να κάνουν για να την οικονομία. Μια από αυτά τα θέματα είναι κατεξοχήν εθνική αρμοδιότητα. Έχουμε λοιπόν σε αυτή την δέσμη των μέτρων που θα τονώσουν την οικονομία. Προσπαθούμε επομένως όλους τους εμπλεκόμενους να τους συντονίσουμε από πλευρά μας. Πρέπει όντως να αναλυθούν κάποιες ε, πρωτοβουλίες που να βοηθήσουν την της δραστηριότητα των ΜΜΕ. Ήδη κάτι κάναμε και ελπίζουμε ότι κάπως θα βοηθήσουν αυτές μας οι πρωτοβουλίες. Ερώτηση του κύριου Μίτσελ για την οικονομική κρίση, χρηματοπιστωτική κρίση. Κύριε Επίτροπε. Σε αυτή τη στιγμή της χρηματοδοτική κρίσης ε, και ύφεση, ε, η Ευρώπη και τα θεσμικά όργανα της κοινότητας έδειξαν την αποφασιστικότητά του. Ε, είδαμε και το πρόγραμμα οικονομική ανάκαμψη το οποίο παρουσίασε ο κ. Μπαρόζο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πακέτο όσον αφορά τι κρατικέ ενισχύσει επιτρέπεται η χρήση ε, επιταχυμένων διαδικασιών για τις κρατικές, ε, για δημόσιες συμβάσεις και ε, υπάρχει και χορηγείται μια ευελιξία στα κράτη-μέλη σε σχέση και με το έλλειμμά τους μέχρι ότου υπάρξει ανάκαμψη από τη γενικότερη οικονομική κρίση. Το 2007 έγινε μια αναθεώρηση της εσωτερικής αγοράς, η οποία όμως θα πρέπει να συνεχίσει έτσι όπως είχε προβλεφθεί και υπάρχει μια σειρά πρόσφατα υιοθετημένων μέτρων ε, της ε, Κομισιόν που ζητούν την, ε, που, θα, επιφέρουν αν θέλετε την ανάκαμψη και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών θα πρέπει να αναθεωρηθεί το κανονιστικό και ε, πλαίσιο της ε, κοινότητας ε, και το πλαίσιο που αφορά την επίβλεψη και τον έλεγχο κυρίως αναφορά το τραπεζικό σύστημα, την προστασία των καταθετών Νομίζω ότι η άμεση υιοθέτηση των μέτρων αυτών είναι απαραίτητη. Τους επόμενους μήνες η Κομισιό θα, θα εξετάσει ε, ενδελεχώς για το πώς θα μπορούσε να, να θεωρηθεί το κανονιστικό πλαίσιο έτσι ώστε να ε, σε κάποια σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Θα απαιτείται καλύτερη συνεργασία και καλύτερο συντονισμό ε, ανάμεσα στις κρατικές αρχές. Ε, θα πρέπει να αποφύγουμε τον προστατευτισμό. Θα πρέπει να περιοριστεί το κόστος ε, των κεφαλαίων. χρειάζεται μια κάποια ευελιξία. Αυτό, αυτή όμως η ευελιξία δεν πρέπει να οδηγήσει σε παραβίαση των αρχών που διέπουν την εσωτερική αγορά. δεν θα πρέπει να παραβιάσουμε τις αρχές της ε, εσωτερικής αγοράς ούτε τις βασικές, τις ουσιώδεις ελευθερίες και τις αρχές ε, της διαφάνειας και της αναλογικότητας. Θα πρέπει να υπάρξει μια ισότητα, αν θέλετε, αντιμετώπισης η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται και να, η οποία θα πρέπει να διασφαλιστεί έτσι ώστε να ελεγχιστοποιήσουμε τις ε, συνέπειες της ε, χρηματοπιστικής κρίσης ε, στην γενικότερη οικονομία. Οι ερώτησεις Μίτσελ και Κρόουλη θα αντιμετωπιστούν μαζί. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και ότι η φωνή σας κύριε Επίτροπο θα βελτιωθεί λίγο. Σας ευχαριστώ για την απάντηση με χαρά ακούω ότι δεν αναβιώνει ο προστατευτισμός γιατί εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο δεν θα είχαμε ανάκαμψη στην Ευρώπη. Ανάκαμψη στην Ευρώπη θα υπάρξει όμως. Και καλό τον Επίτροπο να αρχίσει να συζητά, συζητεί ακριβώς αυτή την ανάκαμψη. Τα σχόλια που ακούγαμε τον τελευταίο καιρό που μεταδίδονται μάλιστα το σημερινό τύπο σχόλια του Προέδρου Τρισέ που προβλέπει ανάκαμψη το 2010, θα ήθελα ο Επίτροπος να αρχίσει ήδη να τα συζητεί, να συζητεί το μέλλον τώρα, να μην χάνουμε χρόνο και επίσης να εξετάσει και, την, το μέλλον της Ευρώπης ως κύριο ανταγωνιστή πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας επιτρέψω περισσότερο χρόνο. Κύριε Κρόλη, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Επίτροπο για την απάντησή του. Θα έλεγα λίγο ουίσκι μέσα σε ένα ζεστό ποτήρι νερό και δύο σταλιές λεμόνι θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ να γλυκάνει το λαιμό του. Για τα οικονομικά μέτρα ανάκαμψης. Αυτό που βλέπουμε του τελευταίους μήνες ήταν ε, συντονισμένη δράση ως μόνη ανταπόκριση. Η μόνη ανταπόκριση απέναντι στην ε, διεθνή οικονομική κρίση. Ερωτώ λοιπόν, υπάρχουν σχέδια ή αρχικές ε, επαφές ίσως με την ε, νέα κυβέρνηση στις ΗΠΑ, την κυβέρνηση Ομπάμα, για να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα για συντονισμένη δράση και από αυτή την πλευρά. Ο Επίτροπος. Κύριε Μίτσελ ε, είναι βέβαια πολύ αισιόδοξο να λέει ότι δεν είναι απάντηση ο προστατευτισμός διότι ασφαλώς κάποια κρατημέλη θα το βρουν αυτό ως μοναδική ευκαιρία να επαναφέρουν τον προστατευτισμό. Δεν θέλω όμως να απαντήσω τα εξής. Πρώτον πρέπει να επαγρυπνούμε. Εφαρμόζεται σωστά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να πάτε στο οποιαδήποτε μέτρα αντιβαίνουν στην νομοθεσία αυτή. Πρώτον και δεύτερον για τα κράτη-μέλη αυτά λέγω το εξή ότι ο πολίτης πιστεύει ότι τέτοια μέτρα θα παρατείνουν την ε, ε, οικονομική κρίση και την ύφεση ε, όπως είπε και ο κύριος Μίτσελ. Μόνο που δεν συμφωνούν όλοι μαζί μας ασφαλώς και κάποιοι ευρωβουλευτές θα διαφωνούν και με εσάς και με μένα κύριε Μίτσελ. Επίσης δεν θέλω να πω ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να εξισορροπηθεί αυτή η αρνητική επιχειρηματολογία που ακούγεται ως προς την οικονομική κρίση με ρεαλιστικά σχόλια που όποτε θα είναι και υπερβολικά απεσιόδοξα. Διότι δυστυχώς στον κόσμο που ζούμε, είτε εδώ, είτε στα κράτη-μέλη μας, είτε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούγονται και φαίνονται κάποιες διαθέσεις για υπερβολικά αρνητική αξιολόγηση των οικονομικών προβλημάτων. Βεβαίω, πρέπει να εξορροπηθεί ο ρεαλισμός και με τις σωστές οικονομικές προβλέψεις, η ρεαλιστική ισορροπία μεταξύ της απεσιοδοξίας και του ρεαλισμού βεβαίως δεν ξέρω που θα βρεθεί. Γιατί χάρη σε αυτή την ισορροπία θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε την αισιοδοξία. Η αισιοδοξία η οποία είναι ένα, το, μια τόσο λεπτή ισορροπία και που μπορεί να χαθεί μέσα σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να δώσουμε σωστές απαντήσεις και χάρη στα έγγραφά μας και χάρη στις προσπάθειές μας πείθοντας τους πολίτες. Για τον κύριο Κρόρε τώρα και την ερώτησή του ως προς τη δυνατότητα να συζητηθούν τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά αυτά αισθήματα με την, κυβέρνηση των, το, νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Έχουμε Υπάρχει βέβαια στις ΗΠΑ πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, ίσως να είστε ενήμερο που ορίζει το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να πράξει η υπό ανάληψη νέα κυβέρνηση ή μη εγκατασταθεί σε ακόμη νέα κυβέρνηση. Όταν εγκατασταθεί όμως η κυβέρνηση αυτή ασφαλώς θα αναλάβουμε επαφέ. Και άλλωστε έχουμε και από το Διεκτατικό Συμβούλιο όπως ε, την, ε, ε, θέματα που συζητούνται διαρκώς όπως ε, τη Συμφωνία για Οικονομική οικονομικές πράξεις κτλ. Όταν όμως, όταν όμως εγκατασταθεί η νέα κυβέρνηση Ομπάμα θα αναλάβουμε τις επαφές. 54-66 θα λάβουν γραπτές απαντήσεις και τώρα κλείνει η συνεδρία. Θα επανέλθουμε στις 9 το βράδυ. Ευχαριστώ.